Euh, Καλησπέρα. Να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα αρχίσουμε με την έγκριση τη ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν ε, διαφωνίες ή σχόλια, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη ω έχει. Έχετε λάβει επίσης τα πρακτικά της 3ης Δεκεμβρίου 2012 της ε, συνεδρίασής μας. Αν έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτά, παρακαλώ να τα γνωστοποιήσετε στη γραμματεία. Πριν από το τέλος της συνεδρίασής μας, της συνεδρίασής μας ε, εγκρίνονται. Επίσης λάβατε και στο φάκελό σας τις ε, συστάσεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 18 Δεκεμβρίου αν ε, έχετε ε, ε, σχόλια ή παρατηρήσεις πρέπει να τα γνωστοποιήσετε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αλλιώς εγκρίνονται όσα έχουν. Εγώ δεν έχω καμία ανακοίνωση να σας κάνω. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσεις. Ναι, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, έχουμε μία ανακοίνωση σε σχέση με την ανακοίνωση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχα έρθει τον Ιούνιο να σας μιλήσω για τέσσερις μεγάλες ανακοινώσεις που είχαν δρομολογηθεί τότε όσον αφορά τη μετάβαση, την ε, κοινωνική προστασία, την αντοχή και τις ε, ε, οργανώσεις ε, τις αστικές έχουν ε, ολοκληρωθεί ειδικά για την κοινωνική ασφάλιση εγκρίθηκε στα μέσα Αυγούστου του 2012 για τη μετάβαση και την αντοχή εγκρίθηκαν στις 3 Οκτωβρίου και η τέταρτη εγκρίθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου. Εδώ έχουμε τον συνάδελφό μου, τον Wolfgang Στράινερ, ο οποίος θα σας πει ορισμένα πράγματα. Είναι από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Θα σας μιλήσει για την ε, ανακοίνωση για την αντοχή, η οποία είναι πολύ σημαντική και την είχαμε ε, στο μυαλό μας εδώ και πολλά χρόνια. Πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και μία ακόμη ανακοίνωση που θέλουμε να δροχομολογήσουμε, που αφορά τη δουλειά που μπορεί να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε σε αναπτυξιακά θέματα με τις τοπικές αρχές. Σκοπό έχουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερο τη δουλειά των τοπικών αρχών ε, στην επεξεργασία, ε, τον προβληματισμό αλλά και την εκτέλεση, την υλοποίηση όλων αυτών των αναπτυξιακών συμφωνιών που έχουμε με τις χώρες δικαιούχους. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, τον ε, κύριο Βόλφαν Στρέιτερ. Έχετε το λόγο κύριε Στρέιτερ. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σημειώσετε δύο κείμενα που υιοθετήθηκαν. Το πρώτο αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Εθελοντική Ανθρωπιστική Βοήθεια, EU Volunteers, που υιοθετήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου και η Κομισιόν προέβαλε αυτήν την πρωτοβουλία η οποία πηγάζει άμεσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή η η εθελοντική ανθρωπιστική βοήθεια θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και στα ανθρωπιστικά, <clears throat> σε ανθρωπιστικές αρχές ε, και θα συμπεριλαμβάνει την ε, εκπαίδευση εθελοντών ε, οι οποίοι θα υποστηρίζουν ευαίσθητες κοινότητες πολιτών και ε, θα τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις ε, ανάγκες τους και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο αρχίζουν αυτή τη στιγμή και βεβαίως είμαστε λίγαν πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας επί της προτάσεως αυτή ε, εμπίπτει μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και ο στόχος είναι να τεθεί ενισχύ αυτή η πρωτοβουλία 1η Πρώτου 2014. Όσον αφορά την ανακοίνωση αντοχής ε, που είναι ένα κοινό, μια κοινή προσπάθεια ΔΕΒΕ καλύπτει τις ε, τελευταίες μας προσπάθειες, ε, τα πιο επίκαιρα, τις πιο ε, επίκαιρες εξελίξεις στο κέρας της Αφρικής και τονίζει πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις κρίσεις στο σημείο αυτό του κόσμου. Στο τέλος της ανακοίνωσης θα βρείτε τις ενέργειες τις οποίες προγραμματίζουμε να υλοποιήσουμε για να αποφευχθούν οι καταστροφές και, να, και η πρόληψη των καταστροφών σε αυτές τις χώρες και το, το, η ανακοίνωση αυτή αφορά το πρώτο τετράμινο του 2013. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε περνάμε στο πρώτο ε, θέμα της ημερήσιας διάταξή μας, το πρώτο ουσιαστικό θέμα, που αφορά ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την ετήσια έκθεση 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό. Ο κύριος Έντουαρτ Κοζούσνικ είναι ο εισηγητή μας για το σχέδιο γνωμοδότησης. Κύριε Κουζουσνίκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα μετάφραση του κειμένου στα τσέχικα, οπότε έχω μεγάλη επιλογή γλωσσών, αλλά εγώ θα διαλέξω τη γλώσσα του Θερβάντες, την οποία και αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου για την προετοιμασία από όλες σχεδόν τις πολιτικές ομάδες. Ε, κάποιοι έλαβαν σχόλια, ε, ε, απέστειλαν σχόλια, κάποιοι άλλοι όχι και από αυτούς που έστειλαν σχόλια νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Η πρόταση γνωμοδότησης ε, βρίσκεται ενώπιόν σας και θα ήθελα να επισημάνω δύο πολύ σημαντικά σημεία, τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε, διότι τα δύο αυτά σημεία ε, είναι αυτά τα οποία διέπουν όλο μου το υλικό. Καταρχάς έχουμε αυτή τη λεγόμενη soft power, την ήπια δύναμη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η επιρροή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι ε, όλα ένα και ισχυρότερη κάθε χρόνο, ε, χάρη σε αποστολές παρατήρησης εκλογών και εντατικοποίηση των προσπαθειών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από πλευράς μου όμως θα πρέπει να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, ώστε τα αποτελέσματα μας σε κάποιες περιπτώσεις να μην μείνουν μόνο συζητήσεις για την πέμπτη το βράδυ, το απόγευμα στο Στρασβούργο. Το δεύτερο ισχυρό σημείο είναι η αποτελεσματικότητα των κονδυλίων που εγκρίνονται, ιδίω εν καιρό κρίση ε, όπως βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εάν ε, επενδύσουμε οικονομικούς πόρους ε, σε κάποιες από αυτές τις περιοχές θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις και τις διάφορες οργανώσεις πρωτίστως αποτελέσματα, τα αποτελέσματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί και διαφάνεια. Είμαι ε, ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις, είμαι ανοιχτός προς συζήτηση και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ όλους. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι, αν θέλετε να πάρετε το λόγο για τη γνωμοδότηση αυτή. Κύριε Σφένσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για μια εξαιρετική γνωμοδότηση. Είμαι σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ και δεν έχουμε να προσθέσω πολλά σε αυτά που ήδη ελέγχθησαν. Ίσως στην παράγραφο 2 θα μπορούσαμε να αναφέρουμε επίσης και το, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ενίσχυση της Δημοκρατίας, το EED. Και θα υποβάλω μερικές ε, ε, μικρές τροπολογίες, σύντομες τροπολογίες για να βελτιωθεί το κείμενο, αλλά γενικά πιστεύω ότι το σχέδιο γνωμοδότηση είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Είναι εδώ, είναι εδώ ο κύριος Μίκαλης Φαν. Ωραία, να δώσω τώρα ε, τότε στον Αλεσάνδρο Βαλτιμπρίνε, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο. Ούτε εκείνο έχει έρθει. Α, εδώ είστε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα σχόλιά του και τον ειδικό εισηγητή επίσης για τα σχόλιά τους. Εκπροσωπώντας την Κομισιόν θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι το σημείο 2 των προτάσεων που προβλέπει την ενίσχυση ε, της υπηρεσίας για την ενδυνάμωση της δημοκρατίας ε, διεθνώς ε, είναι <clears throat> σωστό. Υπάρχει ακριβώς ο νέος κανονισμός για το EAD και ο στόχος της Κομισιόν είναι να υποστηρίξουμε περαιτέρω οργανισμούς, ιδρύματα και υπηρεσίες οι οποίες εργάζονται προς αυτό το σκοπό ε, για να μπορέσει η βοήθεια την οποία χορηγούμε να χρησιμοποιείται κατά το βέλτιστο τρόπο, πιο ενεργά κλπ. Ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν και στους κύκλους της Κομισιόν γίνεται μια συναφή συζήτηση και διαβλέπω από την πλευρά της Κομισιόν ότι η συζήτηση είναι ικανοποιητική όσον αφορά τη βάση αυτή για την έξεση, τη, γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάνη ήρθε? Όχι. Καλά. Σας υπενθυμίζω τότε ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για τη γνωμοδότηση αυτή είναι 11 Οκτωβρίου. Ίσως και ο κύριος Κοζούσνικ θέλει να ξαναπάρει το λόγο για να συνοψίσει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε τις ε, προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών. Μπορούμε να τις επεξεργαστούμε και στη συνέχεια να ετοιμάσουμε την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Le prochain... Μάλιστα, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μα είναι το 8. Στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το κέρα τη Αφρική. Η αντιπρόεδρό μα, κυρία Στρίφλερ, είναι η εισηγήτριά μα. Πριν της δώσω το λόγο όμως, θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της πρεσβείας της Αιθιοπίας που ήρθαν να παρακολουθήσουν αυτό το σημείο της ημερήσιας διαταξή μας και ειδικότερα τον κύριο Τεφέρι Ντέστα που είναι ο ε, βασικός ε, ε, πρόξενος. Κυρία Στρίφα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κέρας Αφρικής. Γνωρίζετε ότι υπάρχει δέσμευση της Ευρωπαϊκής, Επιτροπή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκύπτει από τη σημασία τη γεωστρατηγική της περιοχής, των, στις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολύ καιρό με τις χώρες της ε, περιοχής αυτής και την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, συνεχίσει να καταπολεμά τη φτώχεια στις περιοχές αυτές για να μπορούν να έχουν οικονομική αυτονομία. Τα τελευταία 50 χρόνια η περιοχή έχει ε, δει ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερη πολιτική αναστάτωση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υποστηρίξει τους πληθυσμούς της περιοχής για να ενισχύσει την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ευημερία και να ευαισθητοποιήσει τις κυβερνήσεις ε, ως προς την ευθύνη τους. Στις 14 ε, Νοεμβρίου 2011 ε, οι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν ένα έγγραφο το οποίο ε, δείχνει τα μέσα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, τα στρατηγικά μέσα που έχει στη διάθεσή της σε εταιρική σχέση με την, Αφρικανική Ένωση και με τους βασικούς διεθνείς εταίρους. Πέντε προτεραιότητες θέτει για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, πολιτικές δομές σταθερές που μπορούν να αποκριθούν στη στρατηγική αυτή, πρόληψη και αντιμετώπιση των κρίσεων, άμβλυνση των απειλών που προέρχονται ε, από την περιοχή και που απειλούν την ασφάλεια και επίσης ενίσχυση των ε, προσπαθειών ε, ε, οικονομικής ανάπτυξης, καταπολέμησης της φτώχειας και επίσης ε, οικονομική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Για το συντονισμό των προσπαθειών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2012 έχει έναν ειδικό εκπρόσωπο για το κέρας Αφρικής, ε, ο κύριος Αλεξάνδρε Ρόντος, ο οποίος επικεντρώθηκε στη Σομαλία σε πρώτη φάση, λόγω των συγκρούσεων που υπάρχουν εκεί και λόγω των φαινομένων πειρατών ε, στην ευρύτερη περιοχή. Ε, σας υπενθυμίζω την ε, έγκριση του σχεδίου δράσης που σκοπό έχει να αποκρισταλώσει καλύτερα τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα ήταν πολύ κατακαιρματισμένη η δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορα μέσα. Μετά από ένα χρόνο όμως δεν υπάρχει καμία απολύτως βελτίωση ως προς αυτό. Θα ήθελα να χαιρετήσω ε, τη νέα στρατηγική που ανέπτυξε το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κέρας Αφρικής και που σκοπό έχει να κλείσει το φαύλο κύκλο ε, της ε, πολιτικής αναστάτωσης στην περιοχή. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια στενή συνεργασία μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, όπως επίσης και να ενισχύσει την αντοχή των κρατών και των πληθυσμών για τις μελλοντικέ κρίσεις. Θα ήθελα να ζητήσω η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ενισχύσει τις επιμενικές κοινότητες της ε, περιοχής γιατί είναι ένας βασικός τρόπος ε, συνεργασίας, συντονισμού όπως επίσης και για να συνδεθεί η ανάπτυξη με την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι δύσκολο να δούμε ακόμη τι συνέπειε τη προσπάθεια αυτή. Επίσης, η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητα και η καταπολέμηση της ε, πειρατεία και της ε, τρομοκρατίας ε, δεν πρέπει να εξαφανίζουν το βασικό στόχο που είναι η καταπολέμηση της φτώχειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ε, σκοπό έχει αυτό το συνδυασμό μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της οικονομικής ανάπτυξης και επειδή πρωτοστατεί στην περιοχή θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για την ε, εξάλληψη της φτώχειας ε, που είναι ενδυμικό φαινόμενο όπως επίσης και τα φαινόμενα αναρχίας που διαπιστώνονται στην περιοχή. Δεν θα μπορούσαμε επίσης να δούμε τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει η κατάσταση το κέρας αφαιτής για τις περιοχές της τις κοντινές όπως για παράδειγμα την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ. Λόγος τώρα σε εσά συνάδελφοι, ε, αν θέλετε να ανταλλάξετε απόψεις με την κυρία Στρίφλερ. Αν όχι, δίνετε το λόγο, δίνω το λόγο ε, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, τον κύριο Ντίτμαρ Κρίσλερ, για να σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στη συζήτηση σας. Είμαι αναπληρωτή επικεφαλή του τμήματο ε, Γεωγραφικού Καταμερισμού στην Εξωτερική Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, για το κέρα τη Αφρική. Η γνωμοδότηση τη ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει την αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου για το κέρα τη Αφρική συμμετέχουν ενεργά οι ειδικοί εκφρέσεις ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για το κέρας Αφρικής και για το Νότιο Σουδάν και το Σουδάν. Θα υποβληθεί ε, τον επόμενο μήνα η γνωμοδότηση για να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης. Η εξάλληψη της ένδειας είναι ένας από τους σημαντικούς στόχους αυτού του στρατηγικού πλαισίου. Το στρατηγικό πλαίσιο αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις της ανάπτυξης συνδέονται στενά με θέματα ασφαλείας, και με άλλα λόγια πιστεύουμε ότι το να επιτύχουμε ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια είναι θεμελιώδη σημασία προκειμένου να μειώσουμε την ένδυα. Ε, γι' αυτό το στρατηγικό πλαίσιο καθορίζει μια συνολική προσέγγιση η οποία ε, καθορίζει όλες τις πολιτικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της, ε, κυρίως οικονομικά, πολιτικά όργανα και όργανα ασφαλείας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα αίτια της σύγκρουσης και τα στοιχεία τα οποία αποτελούν πρόσκομα στην ανάπτυξη. Η πρόσφατη, ε, η φέρπουσα συγγνώμη, σύγκρουση μεταξύ ε, Αιθιοπίας και Ερυθρέας ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δυναμητήσει την κατάσταση σε όλη την περιοχή και έχουν ήδη αναλυφθεί οι δράσεις προκειμένου να υπάρξει ενεργό συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό μπορεί να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή της ε, συμφωνίας που έγινε στο Αλγέρι. Η κατάσταση στη Σομαλία επίσης αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Εδώ καλωσορίζουμε τα, ε, ε, την ειρηνική ολοκλήρωση της 10 ε, Σεπτεμβρίου της κατάστασης στη Σομαλία, γεγονός το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε μια ειρηνική κατάσταση στη Σομαλία και ε, επιδοκιμάζουμε επίση και το διορισμό του νέου Πρωθυπουργού και ελπίζουμε να σχηματιστεί το συντομότερο δυνατόν κυβέρνηση. Για αυτή τη νέα κυβέρνηση στη Σομαλία θα πρέπει ε, ε, καθήκον να είναι να εδρώσει, την επιτυχία της συμφωνίας, να υπάρξει συμφιλίωση και να ανασυσταθούν οι νέε πολιτικέ δομάς. Η νέα ε, κυβέρνηση της Ομαλία θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει διαφάνεια όταν θα δίνονται κονδύλια προς όφελος του λαού της. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, από πλευράς ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο νέος ειδικό εκπρόσωπος ε, της Ομαλίας ε, και ο ειδικό εκπρόσωπος ε, για το κέρας της Αφρικής δεσμεύονται να προχωρήσουν τα θέματα αυτά με την ηγεσία της Ομαλίας. Αυτό θα γίνει εντείνοντας την ευρωπαϊκή παρουσία στο Μογκαντήσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστόματος του κυρίου Ντουσαρτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προς το παρόν συμφωνώ με τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και είμαι στη διάθεσή σας αν υπάρχουν περαιτέρω ερωτήσεις. <laughs> Έχετε το λόγο κύριε Στρίφλερ για να συνοψίσετε. Δεν υπάρχει λόγος. Τα σχόλιά σας ευπρόσδεκτα είναι. Αν σκεφτείτε τίποτα άλλο, να μου το πείτε. Σα υπενθυμίζω ότι μέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, 12 ώρα το μεσημέρι, έχετε χρόνο για να καταθέσετε τροπολογίε και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 5 Νοεμβρίου για τη γνωμοδότηση αυτή. Έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα. Ο κύριος Σαλόμ, που είναι υπεύθυνο για το επόμενο θέμα της ημερής διάταξης, δεν έχει έρθει, οπότε πρέπει να πάμε στο 10, που είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Αλφ Βένσον σε σχέση με την αναθεώρηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. αναφέρεται στο θέμα των στρατηγικών που σκοπό έχουν να καταστήσουν πιο αποτελεσματικές και πιο συνεκτικές δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θυμάστε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε αυτήν την έκθεση, να την εξετάζουμε γιατί κάναμε μια πολύ μακρόχρόνια ψηφοφορία ε, για το DCI, για το Μέσο Αναπτυξιακή συνεργασία. Τότε ο κύριος Βένσον ε, είχε την καλοσύνη να αποδεχθεί την ε, αναβολή της έκθεσή του, η έκθεσή του και σήμερα δέχεται ένα τέταρτο πριν να μας την παρουσιάσει. Έχετε το λόγο κύριε Βένσον και σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ εμένα, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη θυσία. Το ζήτημα το οποίο συζητούμε σήμερα αφορά μια πολύ σημαντική στρατηγική. Βρισκόμαστε ενώπιον μια νέα στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρωτοβουλία σα, την οποία επιδοκιμάζω ιδιαίτερα, ε, διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικά φυσικά και για την Επιτροπή μας, αλλά και για όλες τις δραστηριότητες ε, που εξελίσσονται, ε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στο θέμα αυτό σε όλα τα θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός παράγων στο διεθνές προσκήνιο. Είμαστε ίσως ο μόνος ο οποίος προσδίδει τόσο μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά. Για τη νέα αυτή στρατηγική λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι ένα συντονισμό. να μιλούμε με ε, πιο στεναρή φωνή. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ε, πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία. Περιλαμβάνει πάρα πολύ καλές ιδέες και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδης ελευθερία είναι πολύ σημαντικές πτυχές ε, και πολύ σημαντικά στοιχεία διαπραγμάτευσης ε, στην πολιτική διεθνούς ασφαλείας. Το θεματολόγιο λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και εμείς ε, να συμμετέχουμε στα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. θα πρέπει να γίνει μια πολύ καλή αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπινών δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες ε, οι οποίες λαμβάνουν ε, ε, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και μια παράγραφος η οποία αναφέρεται στη σημασία μιας συνεκτικής αξιολόγησης για να μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι κάποια ανθρώπινα δικαιώματα θα βελτιώσουν την κατάσταση στις χώρες τουλάχιστον που βοηθούμε. Θα πρέπει επίσης να εγγυηθούμε ότι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ποτέ δεν θα πρέπει να ε, μεταφραστεί σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνοχή στην πολιτική ανάπτυξη ε, και αυτό για μένα είναι υψή τη σημασία. Όπω σα είπα και προηγουμένω, θα ήθελα να επιμείνω ε, στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη θεμελιώδη ελευθερία. Παρουσιάστηκαν αρκετέ τροπολογίε, τι οποίε ε, στο μεγαλύτερο βαθμό του θα υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ στου συναδέλφου λοιπόν που κατέθεσαν τροπολογίε και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η ΕΕΔ έχει το λόγο τώρα. Ο κύριος Φαν. Είστε πολύ καλή, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι μετά από την εξέταση των προτάσεων του εισηγητή είναι πολύ δύσκολο να διατυπώσω οποιαδήποτε αντίρρηση. Απλώς θα ήθελα να σχολιάσω δύο σημεία, δύο σημεία που έθιξε. Το πρώτο αφορά την αξιολόγηση, ιδίω στα πλαίσια της στήριξη του προϋπολογισμού και επιβεβαιώνω ότι αυτό ήδη τρέχει, ήδη συμβαίνει. Ε, τους τελευταίους μήνες επεξεργαζόμαστε ένα νέο μηχανισμό και τον επεξεργάζεται η Διαρκής Επιτροπή Στήριξης του Προϋπολογισμού και έτσι ε, θα ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές αυτού του νέου μηχανισμού στις αποφάσεις που θα ληφθούν και θα λαμβάνονται. Δεύτερον, ε, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό καλύπτεται ασφαλώς μέσα στο πρόγραμμα δράσης που συνοδεύει το στρατηγικό πλαίσιο, όπου αναφέρεται ρητά ότι κατά πρώτο και κύριο λόγο θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις μελέτες επιπτώσεων και επιβεβαιώνω ότι και αυτό εφαρμόζεται από την Κομισιόν. Οπότε με την άδειά σας θα σταματήσω εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκπρόσωπο τον κύριων Βάλτον Μπριντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο θα θέλαμε και εμείς να υποστηρίξουμε τις προτάσεις του κυρίου Σβένσον και όπως είπε και ο συνάδελφός μου από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφισβητήσει ή να διαφωνήσει με κάτι που αναφέρει. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που στο σημείο 7 αναφέρει μια νέα προσπάθεια υποστήριξης των ατόμων που ε, υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγματι, αυτή ήταν μία ιδέα την οποία παρουσίασε η Κομισιόν για τον νέο κανονισμό και προτείναμε να ε, αυξηθεί ο κανονισμός ακριβώς για να προβλεφθεί ε, τα αναγκαία κονδύλια προστασίας και ενίσχυσης ε, των ακτιβιστών που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω το σημείο 5 που λέει ότι θα πρέπει να σηματοθούν στρατηγικές των χωρών και τον ευνοήσει στον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των ενισχύσεων προς τρίτες χώρες. Αυτό είναι κάτι που ελπίζουμε να γίνει βεβαίω σε συντονισμό με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αλλά ήδη τώρα ε, με, το, με τις νέες προτάσεις για την υπηρεσία υποστήριξη της δημοκρατίας και το νέο πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήδη η Κομισιόν αναθεωρεί και μελετά τη στρατηγική των τρίτων χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δηλαδή μια ε, ενέργεια, μια στρατηγική η οποία ήδη εφαρμόζεται και είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 20 Σεπτεμβρίου είχαμε θέση ως ε, ημερομηνία υποβολής τροπολογιών γιατί λέγαμε να ψηφίσουμε αύριο τη γνωμοδότηση αυτή. Αύριο λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε την ε, ε, γνωμοδότηση του κύριου Σβέντσον. Θέλετε να την ψηφίσουμε αύριο, την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για τα θετικά σχόλια. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε συνεχώς την τρέχουσα κατάσταση όταν συζητούμε για, τις ανθρώπινες, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ως αυτονόητο ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί κάποτε θα συνεχίσουν να ισχύουν ε, εσαΐ. Ε, είναι σημαντικό να εξετάζουμε συνέχεια τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίζεται η ακαιρεότητα του ατόμου παντού και πάντοτε. Άρα θα ψηφίσουμε αύριο τη γνωμοδότηση αυτή. Ο κύριος Ντέσπεργ μήπως είναι εδώ. Α, είστε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε πίσω τότε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξής μας, την έκθεση για την ειδική ε, έκθεση που αφορά την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για ε, στην αναπτυξιακή της βοήθεια και την επισητιστική ασφάλεια στην υποσαχάρη Αφρική. Θα ακούσουμε την άποψη του Ενρίκη Γκερέρο Σαλόμ για την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επισητιστική βοήθεια στην Υποσαχάρη Αφρική. Πρόκειται για μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής του 2011. Η αρμόδια ε, επιτροπή είναι η Επιτροπή ελέγχου του προπολογισμού. Για την ανταλλαγή απόψεων έχουμε εδώ ε, τον κύριο Βέσπεργ ε, που είναι ε, το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου που είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό στο ελεγκτικό συνέδριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βέσπεργ για την παρουσία και σας δίνω το λόγο ευθύς αμέσως. Thank um, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω ε, σύντομα ε, τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα αυτής της ε, έκθεσης για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και την επιστημιστική ασφάλεια. Καταρχήν, επισητιστική ασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι να υποφέρουν από πείνα. Και είναι μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι ανα πάσα στιγμή στερούνται την επαρκή πρόσβαση σε, σε σύντηση και στις πηγές της παραγωγής τροφίμων η επιστημιστική ασφάλεια είναι ένα καυτό πρόβλημα στην υποσαχάρη Αφρική όπου 239 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή 30% του συνολικού πληθυσμού υποφέρουν από πείνα. Από το 2002 μέχρι το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξασφάλιση της επισητιστικής βοήθειας στην Ποσαχάρη Αφρική, της επισητιστικής ε, ασφάλειας και αυτό έγινε μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας με, με μονομένες χώρες της υποσαχάρης Αφρικής αλλά και μέσω των διαφόρων μέσων υπηρεσιών και ε, ε, ε, διευκολύνσεων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε πολλά προγράμματα διάθεσης, ε, βραχυπρόθεσμης διάθεσης ε, μέσω σιτισμού και επισητιστικών προϊόντων για επίσης σπόρους που είναι αναγκαίους και άλλα μέσα αναγκαία για την καλλιέργεια τροφίμων και παραγωγή τροφίμων. Υποστηρίξαμε επίσης προγράμματα <coughs> έρευνας και τεχνολογίας στον γεωργικό τομέα ε, ώστε να ισχυθούν οι εθνικοί πόροι που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Το 2008 αναπτύξαμε μία ε, δύναμη άμεσης δράσης η οποία να μπορεί να επέμβει όταν θα έβλεπε να αυξάνονται κατακόρυφα οι τιμές των τροφίμων στις χώρες αυτές. Τώρα λίγα λόγια για την ελεγκτική εργασία την οποία επιτελέσαμε. Το ελεγκτικό συνέδριο εξετάζει αν η βοήθεια, η επιστημιστική βοήθεια είναι αποτελεσματική στην υποσαχάρη Αφρική. Εάν η ευρωπαϊκή επιστημιστική βοήθεια έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες της χώρας στην οποία διατίθεται και αν οι παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές, όπως είπα. Εμείς ε, ελέγχουμε τις τρεις πτυχές της επιστημιστικής ασφάλειας. Διάθεση, πρόσβαση και χρήση των προϊόντων σύντησης. Μαλάβια and Rwanda. A further in-depth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 to the development of incoming earning capacities of the beneficiaries. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στον ε, κύριο Γκερέρο Σαλόμ για να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του. Sí, muchas gracias. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Βέσπερκ, μέλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Μόλις ακούσαμε και τις ε, βασικές γραμμές της ε, έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχουν τρεις σημαντικές ερωτήσεις που γίνονται εδώ. Η πρώτη είναι εάν η βοήθεια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των τριών μέσων που επισημάνθηκαν ήταν αποτελεσματικοί. Εάν δηλαδή τηρήθηκαν οι στόχοι οι οποίοι είχαν ε, προταθεί, εάν υπήρχε βοήθεια σχετική με αυτό που έπρεπε να συνεισφέρει, δηλαδή εάν συνεισέφερε στη βελτίωση της ε, επισητιστικής κατάστασης ε, αρκετών χωρών, για, τους, για τις οποίες έγινε μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη, και εάν εν Εάν επιτεύθηκαν οι στόχοι οι οποίοι προτάθηκαν, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η στόχη είναι βιώσιμη. Δηλαδή, ότι η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνεχίσει προς ε, αυτή την κατεύθυνση με ε, βιώσιμο τρόπο. Το συμπέρασμα της έκθεσης είναι ε, ότι απαντάει καταφατικά και στα τρία ερωτήματα. Ναι, ήταν αποτελεσματική, ναι, ήταν σχετική αυτή η βοήθεια και σίγουρα μπορεί να είναι βιώσιμη. Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι υπάρχουν και πρόσθετες δυνατότητες από αυτές που έχουν ε, γίνει μέχρι τώρα. Καταρχάς, η δυνατότητα να διαβρινθεί βοήθεια και σε άλλες χώρες, ώστε αυτό που ήταν μια συγκυριακή δράση μέσω του facility να μπορέσει να γίνει πλέον διαρθρωτική δράση και δεύτερον να δοθεί περισσότερη έμφαση ε, στις ε, καθαρά διατροφικές πτυχές. Τέλος, η έκθεση συστήνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μια σειρά από μέτρα Κάποια μέτρα αφορούν ε, το ε, περιεχόμενο της βοήθειας και κάποια αφορούν ε, τη μέθοδο αξιολόγησης για να συμπεριληφθούν και δείκτες εισοδήματος. Εάν περιοριστούμε λοιπόν αποκλειστικά και μόνον στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι ε, ότι είναι αποτελεσματική η βοήθειά μας και ότι είναι σύμφωνη με τους στόχους που έχουμε θέσει. Εάν όμως δούμε τον πραγματικό κόσμο, αν δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στην υποσαχάρη Αφρική, νομίζω ότι η ανησυχία μας ε, θα πρέπει να αυξηθεί παρά το γεγονός ότι η ικανοποίησή μας για τη δράση μας είναι αρκετά ε, καλή. Και γιατί θα πρέπει να ε, μην νιώθουμε ικανοποιημένοι και να ανησυχούμε. Καταρχάς γιατί οι επισητιστικές κρίσεις ε, είναι όλο ένα και πιο συχνές. Και επειδή ακριβώς είναι πιο συχνές, εξορισμού είναι και πιο οξύες. Διότι είναι κρίσεις οι οποίες ε, έρχονται στη συνέχεια προηγούμενων κρίσεων και επομένω επιδεινώνουν κι άλλο την πραγματικότητα εκατομμύριων ανθρώπων που ούτω ή άλλω έχουν πληχθεί και στο παρελθόν από άλλε επιστημιστικέ κρίσει. Υπάρχουν τρία βασικά αίτια ε, για τα οποία ε, πάσχουμε από συνεχείς κρίσεις. Καταρχάς, ε, τα φυσικά αίτια, τα λέμε φυσικά για να κατανοήσουμε αλλήλους, γιατί στην πραγματικότητα προκαλούνται από την ανθρώπινη δράση, δηλαδή σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος και με τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Κάποια άλλα αίτια έχουν σχέση με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση παγκοσμίω, η οποία ε, πλήττει ε, ακόμα περισσότερο τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και κάποια αίτια προέρχονται από κάποια χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς της κοινωνίας τον τρόπο, για παράδειγμα, ε, παραγωγής, τον κυρίαρχο τρόπο παραγωγής. Πρόκειται για ε, κερδοσκοπικές δραστηριότητες ε, που έχουν στόχο μόνο ωφέλη στις τιμές των προϊόντων και επομένως υπάρχουν πτώσεις έλλειψης τροφίμων και κάποιες άλλες έλλειψης προσφοράς προϊόντων σε κάποιες περιοχές του κόσμου. Το συμπέρασμα λοιπόν στο οποίο κατέληξε η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το 2010 για τους στόχους της χιλιακίας ε, είναι ότι ε, απομακρυνόμαστε βαθμιδών από την τήρηση των στόχων. Ε, στην αρχή, το 2000, ε, θεωρούσαμε ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε ένα ουσιαστικό τμήμα αυτών των δεσμεύσεων και τώρα ε, στη σήμερα ημέρα απομακρυνόμαστε για λόγους του οποίους γνωρίζει πολύ καλά η Επιτροπή μας εδώ και δεν θα επιμείνω από αυτόν, αλλά σε μεγάλο βαθμό γιατί η βοήθεια και η συνεργασία για την ανάπτυξη περιορίστηκε σημαντικά ε, σε αρκετά μέρη του κόσμου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και ο βασικός στόχος της εξάλληψης της ε, πείνας ε, εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί και πόρα απέχουμε από την υλοποίησή του. Τώρα, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μας αποστέλει ως μήνυμα, ως ένα από τα βασικά μηνύματα, είναι ότι η απάντησή μας από, μέσα από μηχανισμούς ε, κατεπίγουσας ανάγκης και συγκυριακούς θα πρέπει να γίνουν ε, διαρθρωτικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί ε, πρόληψης ε, της κατάστασης. Η περιγραφή που σας έκανα αυτή τη στιγμή είναι η βάση της γνωμοδότησης που θα σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει πολλά από τα σημεία τα οποία κατ' έχει θίξει εδώ η Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, υπάρχει και η θέση της Επιτροπής Ανάπτυξης ε, σε αρκετές εκθέσεις. Μεταξύ αυτών έχουμε και την ανάγκη να υπάρχουν ε, συστήματα πρόληψης για να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε οξύες επιστημιστικές κρίσεις και όπως είπε και ο κύριος Βάισμπεργκ η θέση και η δράση τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτού του κινδύνου ε, οξείας κρίσης και επίσης ε, συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ε, εντείνουμε τις ε, διατροφικές πτυχές και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει και μία έκθεση για την πτυχή αυτή. Επίσης, ζητάμε να μην ε, παρατηθούμε ενώπιον της διακύμασης των τιμών και την κερδοσκοπία που αντιμετωπίζουμε στην αγορά ε, διατροφικών προϊόντων και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτίστως να προσπαθήσει να βρει μέτρα και ε, στο ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο. Στο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ένας παγκόσμιος παράγοντας που θα μπορεί να ελέγχει ε, τις, αλλαγές, ε, τις αγορές τροφίμων, δηλαδή να τις ρυθμίσει, όχι να τις ε, προστατεύει και επίσης να δημιουργήσουμε και αποθεματικό τροφίμων τα οποία θα αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην κερδοσκοπία. Επίσης, Θέλουμε να ενισχύσουμε την πρόσβαση σε πίστοση σε μικρομεσαίους γεωργούς και φυσικά να επαναλάβουμε τη θέση της Επιτροπής μας ε, υπέρ της συνοχής ε, στις πολιτικές ανάπτυξης. Τέλος, ε, θα ήθελα να παρουσιάσω και μία σκέψη που θεωρώ ότι ο πλειοψηφία, αν όχι όλα τα μέλη της Επιτροπής, θα συμφωνήσει. Βρισκόμαστε εν μέσω της συζήτησης για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν τρεις ομάδες χωρών στο Συμβούλιο. Μία ομάδα η οποία είναι υπέρ ε, της αύξησης ε, του συνολικού ε, ποσού των δημοσιονομικών προοπτικών για τις πολίτες προοπτικές και το ίδιο έχει ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 5% αύξηση για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει επίσης μια άλλη ομάδα χωρών η οποία είναι υπέρ του να ε, παγώσουμε το ποσοστό και να μείνουμε στους στόχους του 2013 και να είναι οι ίδιοι οι στόχοι στις ε, δημοσιονομικές προοπτικές, που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θα έχουμε μείωση, διότι αν παγώσουν ε, τα κονδύλια για τα επόμενα χρόνια, σημαίνει ότι θα υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες και επομένως δεν θα παγώσουν οι τιμές, αλλά θα μειωθούν. Και τέλος έχουμε και ένα περιορισμό. Εμείς από την Επιτροπή Ανάπτυξης θα πρέπει να κάνουμε δύο αιτήματα. Ε, ένα υπέρ πολιετών ε, δημοσιονομικών προοπτικών ε, οι οποίες θα είναι αυξημένες και δεύτερον, οποιοδήποτε αποτελέσματα και να έχουμε, να μην γίνει τίποτα εις βάρος της ε, αναπτυξιακής πολιτικής. πολλές χώρες, η χώρα μου επίσης, ε, αντιμετωπίζει προβλήματα. Υπήρχαν πολλές αποφάσεις οι οποίες ε, αμφισβήτησαν την ε, σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Ισπανία ε, αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη πλέον έχει επανέλθει στα ποσοστά και στις, στα κονδύλια που είχαμε πριν από μία δεκαετία. Και εδώ θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να υψώσουμε λάβαρο υπέρ της αύξησης ή τουλάχιστον να παραμείνουμε στο ίδιο ποσό, διότι αν συμβεί το αντίθετο δεν θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας, κάτι το οποίο εμείς ε, στην Επιτροπή μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γεροσαλόμ. Ο κύριος Νόησερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ειδική αυτή έκθεση, την οποία μπορέσουμε να δούμε, να κοιτάξουμε και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μία, ένα input, ένα περιεχόμενο που προσφέραμε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω, να κάνω μερικά σχόλια για τους στόχους μετά το 2015. Επειδή μιλάμε για την εξάλληψη της φτώχειας, θα πρέπει να προσεγγίσουμε περισσότερο τα αίτια της φτώχειας παγκοσμίω. Πιστεύω ότι οι στόχοι της ε, χιλιετίας... Βένον καλός όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, φτώχειας, αλλά εμείς προσπαθούμε να γιατρέψουμε τα συμπτώματα. Η φτώχεια αυξάνεται, το φαινόμενο της υποανάπτυξης διατηρείται και η συζήτηση των εξελίξεων μετά το 2015 ξεκινάει για το πώς ε, θα υλοποιηθούν οι στόχοι της χιλιετίας και γι' αυτό ο χρόνος πλησιάζει και θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ πιο έντονα τις επιπτώσεις στις ε, χώρες αυτές που θίγονται και να δούμε τι δυνατότητες ε, συμμετοχής και συνεργασίας υπάρχουν. Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κατανομής των βαρών στις χώρες αυτές οι χώρες της Πασαχάριας Αφρικής είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες, όμως τα δύο τρίτα όλων των ανθρώπων παγκοσμίω που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ζουν σε αυτές τις χώρες. Ε, από αυτό φαίνεται η σοβαρότητα της κατάστασης. Ο συνάδελφός μου, Νέστο, ε, Βάιλερ έχει θέσει ε, στόχους πέραν από τους μετριόφρονες στόχους που είχαμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω μερικά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και ο κύριος Γερέρος Σαλών μας είπε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πέτυχε το στόχο της ε, σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούμε όμως να ξεχνούμε και τις ε, παρενέργειες ε, της, της κοινή γεωργικής και αλληλευτικής πολιτικής ε, που κατέστρεψε ε, γεωργικούς και αλληλευτικούς πόρους της ε, Αφρικής και ειδικότερα σε, περι, σε περιόδους περικοπής που θα μειωθεί η βοήθεια και ενδεχομένως το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι η αλληλευτική πολιτική την οποία αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε και για την οποία κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία μεταξύ άλλων δεν συμφωνούν για τον περιορισμό της ε, αλίευσης ε, στο μέγιστο που μπορούν να αντέξουν οι αλλιευτικοί ε, πόροι, τα είδη που Και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό όταν οι στόλοι μας αλλιεύουν στα αφρικανικά ύδατα. Υπάρχει μια υποκρισία απαράδεκτη την οποία οποία, το γεγονός δηλαδή ότι οι χώρες μας δεν δέχονται να μειώσουν την ε, αλληλεία ε, προς όφελος των ε, παράκτιων πληθυσμών και για οικολογικούς καθαρά λόγους θα μπορούσαμε να μην μειώσουμε τουλάχιστον τη βοήθειά μας προς τις χώρες αυτές όταν έχουμε ε, αλλιεύσει ε, τόσα πολλά είδη στις ε, χώρες αυτές. Το ίδιο ισχύει για το, για το εμπόριο και για τη γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους συναδέλφους που ε, έχουν κάτι να πούν στη χώρα τους, ε, να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η, γεωργική και αληφτική πολιτική μας ε, να είναι 100% υπεύθυνη όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. και να θυσιάσουμε το βραχυπρόθεσμο εμπορικό μας συμφέρον για ένα ε, ευρύτερο συμφέρον των πληθυσμών της υποσαχάριας Αφρικής, ώστε να μπορούν με τις δικούς τους πόρους ε, να τρέφονται οι πληθυσμοί αυτοί. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστόματος του Ζων Πιεραλκιά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μας ε, σε σχέση με την έκθεση ε, για την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που αφορά την επιστημιστική βοήθεια της υποσαχάριας Αφρικής, στην υποσαχάρια Αφρική. Το Ελεκτικό Συνέδριο έκανε καλή δουλειά και εκτιμήσαμε ιδιαίτερα τις επαφές που είχαμε για τη συζήτηση της ουσίας των πραγμάτων, ε, των διαπιστώσεών τους, των πορισμάτων τους και των συμπερασμάτων τους. Για τις βασικές ε, συστάσεις μπορώ να πω ότι έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η οποία δεν διαφωνεί με το να μεταφραστούν αυτές ε, οι συστάσεις σε πράξη, ειδικότερα εν ώψη του προγραμματισμού 2014-2020. Να σας πω ένα παράδειγμα. 52 χώρες εντοπίσαμε, στις οποίες, στις οποίες υπάρχει χρόνια ε, επισητιστική ανασφάλεια, έλλειψη ασφάλειας και ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις ε, αντιπροσωπείες ε, να προβούν σε ένα διάλογο με τις χώρες εταίρους για να δούμε όχι μόνο να, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έλλειψης ασφάλειας, αλλά και πώς μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερους ε, πόρους ε, για να εξαλείψουμε τους στόχους αυτής της, τους, ε, συγγνώμη, τους λόγους ύπαρξης αυτής της έλλειψης επιστηστικής ε, ασφάλειας. Ε, επίσης θέλουμε να δούμε και την πολιτική πτυχή και να την επεξεργαστούμε. Όπως γνωρίζετε στις 3 Οκτωβρίου, την περασμένη Τετάρτη δηλαδή, εγκρίναμε στην Επιτροπή μία ανακοίνωση για την αντοχή ε, με τον τίτλο ε, «Πώς μαθαίνει κανείς από τις επιστηστικές κρίσεις» και πώς βελτιώνεται η αντοχή. Προσπαθήσαμε λοιπόν δηλαδή βάσει των προηγούμενων κρίσεων να δούμε τι μάθημα μπορούμε να πάρουμε. Μεταξύ των προσανατολισμών λοιπόν που προτείνονται στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης υπάρχει και ο στόχος της ε, περαιτέρω ενίσχυσης των ε, ε, ικανοτήτων των χωρών εταίρων να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις και κυρίως τις επισητιστικές. Ένα από τα σημεία που επίσης έθεσε η έκθεση ε, είναι η ε, κακή διατροφή των παιδιών. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ έγκαιρο. Γνωρίζετε ότι αυτό το θέμα υπάρχει εδώ και με μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 2008 όμως μία επιστημονική έκθεση ε, έθεσε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση σε σχέση με το θέμα αυτό της κακής διατροφής των παιδιών 3,5 εκατομμύρια παιδιά τουλάχιστον ε, κάτω από 5 ετών ε, ε, χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω του προβλήματος αυτού. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε στο παρελθόν και το οποίο χρήζει ιδιαίτερη προσοχής από τους, από τους δωρητές. Κάτι ακόμη μεταξύ των 175 εκατομμυρίων παιδιών παγκοσμίω που υποφέρουν από κακή διατροφή διατροφή δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν στο πλήρες δυναμικό τους ε, σωματικής και πνευματική ανάπτυξης. Είναι πήγον λοιπόν να το λύσουμε αυτό το θέμα και για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά και για να επιτρέψουμε σε όλα αυτά τα παιδιά να έχουν το μέλλον που τους αξίζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε όλο ιδιαίτερο για το θέμα αυτό τη ε, κακή διατροφή των ε, παιδιών. Τα κράτη-μέλη έχουν μάλιστα ένα τεχνικό δελτίο για το πώ θα αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και ε, από τη Γενική Διεύθυνση της Ανάπτυξης αλλά και της Ανθρωπιστικής Βοήθειας προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το θέμα για να υπάρξει ένα ε, δελτίο ε, χάραξης πολιτικής για το θέμα αυτό. Μεταξύ των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου για τις δημοσιονομικές Προεπτικές 2014 με 20 υπάρχει το γεγονός, υπάρχει το γεγονός ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον οικονομικό μας κανονισμό για να ε, μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες. Ένας τρόπος ε, να αντιμετωπίσουμε τις επιστηστικές κρίσεις ε, είναι η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της να αντιδράσουν γρήγορα και ουσιαστικά Ε, στην την τελευταία φορά ε, ένα δισεκατομμύριο ευρώ μπορέσαμε να ε, εκταμιεύσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Παρόλα αυτά όμως, δείξαμε λοιπόν την δυνατότητα των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να αντιδράσει. Είπαμε μάλιστα ότι 3 εκατομμύρια δολάρια θα ε, ε, δαπανηθούν ε, στο πλαίσιο αυτό και μάλιστα και στο κέρας Αφρικής το κάναμε. Δείξαμε ευελιξία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη μηχανισμών ευέλικτων, καλύτερα προσαρμοσμένων στην κρίση, στις κρίσεις, γιατί αυτό που κάναμε ως σήμερα για να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιζητιστικών κρίσεων, Μερικές φορές το κάναμε εις βάρος των ε, προσπαθειών ε, που είχαμε καταβάλει για να, δούμε από πού προερχόταν η κρίση αυτή, ποιες ήταν οι αιτίες της κρίσης αυτής. Ε, αυτό λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες χωρίς να μειώσουμε την καταβολή των προσπαθειών για την εξέβρεση των αιτίων της κρίσης. Ελπίζω να απάντησα Είμαι διαθέσιμος και, σε άλλες, ε, και για άλλες ερωτήσεις, αν θέλετε να τις απαντήσω. Συγγνώμη, πρώτη φορά απαντώ ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαι επίσης ε, διαθέσιμος ε, να πω ορισμένα πράγματα και όλες για τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαρίστω να σας βοηθήσω όπως μπορώ. Ευχαριστώ και πάλι, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Βέσπεργ και μετά ο κύριος ε, Γκερέρος Σαλόμ θα πάρει πάλι το λόγο. Ε, θα ήθελα να πω απλώς ότι και εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την συνεργασία που είχαμε με τις υπηρεσίες της Κομισιόν σε αυτή τη φάση. Ο κύριος Γκερέρο έχει το λόγο. Ναι, Ήθελα να πω στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ήδη γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν υπάρχει δεύτερη πρώτη φορά. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν την πρώτη φορά που εμφανίζεστε εδώ στην Επιτροπή, διότι από τη δεύτερη και τρίτη φορά θα δείτε ότι είμαστε λογικοί άνθρωποι όσοι εργαζόμαστε εδώ στην Επιτροπή. Ήθελα απλώς να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο, το οποίο θα αναγράφεται και στη γνωμοδότησή μου στην Επιτροπή Προπολογισμών. Εμείς συμφωνούμε σε μια διαφορετική απάντηση στα προβλήματα της επιστημιστικής ασφάλειας. Ε, ο όρος λοιπόν αυτού του resilience, της αντοχής, ε, είναι και μια ανησυχία που έχουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας συνήθως. Δεν θα πρέπει όμως ε, να εγκαταλείψουμε ολοκληρωτικά τη δυνατότητα να δράσουμε ενώπιον ε, σοβαρών, απρόβλεπτων καταστάσεων ή ε, καταστάσεων που οξύνονται. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η καταστασεων που οξυνονται θεωρω Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει και το ενδεχόμενο είτε να παραμείνει το food facility, το οποίο χρήσιμευσε για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες κρίσεις, ή ένα αντίστοιχο μέσο για τις επόμενες πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Euh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ σημαντική δουλειά της Επιτροπής μας. Και κλεισμένων των θυρών τώρα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων και τις πληροφορίες για τον πρώτο τριμερή διάλογο των ε, άτυπο ε, για το ε, DCI, για το Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Όμως δεν είχε φτάσει η ώρα του σημείου αυτού της ημερήσης διάταξης, γι' αυτό θα διακόψουμε λίγο για 45 λεπτά. Σε 45 λεπτά λοιπόν θα επανέλθουμε και κλεισμένων των θυρών για το τελευταίο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Μετά θα κάνουμε του συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο το πρωί πάλι δημόσια συνεδρίασή μας, 9 η ώρα το πρωί, με την ψηφοφορία. για τα θέματα και κλεισμένα των θυρών μόνο οι συνάδελφοι, οι βοηθοί τους, ε, το προσωπικό των, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το προσωπικό των πολιτικών ομάδων. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλώ να αποχωρήσουν. Διακόπτεται η συνεδρίαση για 45 λεπτά. Μέχρι τις 5 και 4 λέει η Πρόεδρος. Correction, je suspends jusqu'à 5 heures. Nous allons gagner un quart d'heure. Μέχρι τις Πέντε η ώρα διορθώνει ο πρόεδρο, Πέντε η ώρα διορθώνω και όχι πέντε και τέταρτο όπως είπα προηγουμένω. Πέντε η ώρα. Five. Five.